η σύμβαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, ε, θα, θεωρούνται ότι έχουν ισότιμη αξία. Και μιλούμε για μια αμοιβαία αναγνώριση του οικομενικού συστήματος προστασίας ε, των δικαιωμάτων του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένης και της Χάρτας του Τωρίνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πήραμε λοιπόν μία πρόταση ψηφίσματος, ε, ολοκληρώθηκε η συζήτηση και ως εκ τούτου ε, ανακοινώνω το τέλος της συζήτησης. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο το πρωί. Σύμφωνα λοιπόν με την ημερήσια διάταξη έχουμε τώρα τις ε, δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης. Η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, όμως ξεπεράσαμε το χρόνο μας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω όλους όσοι θα παρέμβουν να τηρήσουν αυστηρά το χρόνο που θα τους διατεθεί. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο χώρος της ε, δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ευρωπαϊκός χώρος λοιπόν ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Τα κράτη-μέλη έχουν συνεργαστεί και έχουν εμβαθύνει ιδιαίτερως ε, στη συνεργασία τους σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας, είναι ένα από τα πιο σημαντικά σχέδια που έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εφαρμοστεί σωστά ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι έχουν ενισχυθεί πολύ περισσότερο οι σχέσεις με τον Ευρωπαίο πολίτη. Υπ' αυτή την έννοια ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες πραγματικά νιώθουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να τους ε, δώσει μια προστιθέμενη αξία, έχει να βοηθήσει την, μπορεί να βοηθήσει την καθημερινότητά τους στις πολύ βασικές πτυχές της καθημερινότητάς τους. Ο Ευρωπαίος πολίτης, ας πούμε, μπορεί να απολαμβάνει συνθήκες ασφάλειας, ελευθερίας, δικαιοσύνης και ε, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα επιτέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι γεγονός, αδιαφυσβήτητο. Μάλιστα, ορισμένες αποφάσεις που έχει υιοθετήσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε όλο αυτό το ευρύ πεδίο της δικαιοσύνης και της ασφάλειας και της ε, ελευθερίας στο παρελθόν όταν η συνεργασία ήταν κυρίως ε, μεταξύ των κυβερνήσεων στο πεδίο αυτών αρμοδιοτήτων, ορισμένες αποφάσεις, ε, λέω, έχουν να κάνουν με το θέμα το οποίο συζητούσαμε και προηγουμένως, δηλαδή την ε, διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου, ε, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, εγκλημάτων όπως η γενοκτονία και ούτω καθεξής. Από τον Ιούνιο του 2002 και μάλιστα από τις 8 Μαΐου του 2003, το Συμβούλιο έχει γίνει εξαιρετικά λειτουργικό και έχει υιοθετήσει ε, τα δέοντα ώστε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τη δίωξη ε, των ηθινόντων για τα εγκλήματα αυτά. Θυμόμαστε όλοι, για παράδειγμα, την περίπτωση του Πινοτσέτ. Σε ορισμένες χώρες μέλη ε, αυτή η δυνατότητα έχει ενσωματωθεί και στην εθνική νομοθεσία, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία στην Ισπανία έχουμε τη νομική έννοια της ε, οικουμενικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, ε, για εγκλήματα τα οποία είναι εξαιρετικά σοβαρά, ακόμα και αν έχουν διαπραχθεί εκτός της Ισπανικής επικράτειας, ε, μπορού, μπορεί να υπάρξει άσκηση διώξεων στο εσωτερικό της Ισπανικής επικράτειας, παρόλο που ίσως φαίνεται αυτό ως κάτι το αντιβαίνον επιφανειακά στην τόσο προστατευόμενη αρχή της της ε, εδαφικής ε, ε, χωροθέτησης αν θέλετε του ποινικού αδικήματος. Δηλαδή αυτή η περιβόητη αρχή έχει τεθεί κατά μέρο σε περίπτωση κατά την οποία διαπράττονται εγκλήματα που πραγματικά αποτελούν ένα πολύ βαρύ πλήγμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει αυτό το χώρο δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας στην Ευρώπη και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε το πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης. Η συνθήκη της Λισαβόνας κάνει ε, ο χώρος της ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας να μην είναι μόνο στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και να μην γίνεται μόνο αντικείμενο διακυβερνητικής συνεργασίας, αλλά να είναι πλέον ο χώρος αυτός βασική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχει λοιπόν κοινοτική αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά πλέον και γι' αυτό όλοι χαιρετίζουμε την έγκριση του προγράμματος ε, δράσης της Στοκχόλμης ε, το Δεκέμβριο του 2009 από πλευράς Συμβουλίου. Με το πρόγραμμα δράσης αυτό ε, καθορίζονται συγκεκριμένα καθήκοντα για τα κράτη-μέλη και τα συμφέροντα των πολιτών, η προστασία του Ευρωπαίου πολίτη αποκτούν πλέον υψηλή προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να αναφερθώ και πάλι στη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως για το προηγούμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, με το πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμη, τα κράτη-μέλη πλέον υποχρεούνται να συνεργαστούν με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο προκειμένου να ασκηθούν διώξει και να αποδοθούν ευθύνε για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητα, έτσι ώστε να μην υπάρξει ατιμορρησία. Ε, αφού όλα αυτά έχουν εγκριθεί ε, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Σουηδικής Προεδρίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί, θα πρέπει να υλοποιηθεί, θα πρέπει να μεταφραστεί στην πράξη και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο ε, «Σχέδιο δράσης εφαρμογής του προγράμματος της Στοκχόλμης για την προστασία ε, των πολιτών». Με το πρόγραμμα δράσης λοιπόν της Στοκχόλμης βασιζόμαστε στα προηγούμενα επιτεύγματα και αντιμετωπίζουμε τις νέες προκλήσεις αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες που μας δίνονται με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, ε, Έχουμε λοιπόν ε, πλέον μπει σε μια καινούρια εποχή. Από θεσμικής πλευράς ε, πρόκειται για ένα σημείο επαναστατικό και υπογραμμίζω τη λέξη επαναστατικό. Πρόκειται για μια θεσμική και νομική επανάσταση πλέον και αυτό είναι εξαιρετικά ε, σημαντικό διότι κάτι το οποίο εντασσόταν αμυγός στις αρμοδιότητες κρατών μελών και γινόταν αντικείμενο διακυβερνητικής συνεργασίας πλέον εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής το Συμβούλιο λοιπόν αναγνωρίζει τη σημασία και τον τεράστιο ρόλο που έχει να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης, ως θεσμικός εταίρος ε, στην υιοθέτηση των μέτρων που θα λάβουμε τα επόμενα χρόνια για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Επιτρόπος κυρία Ρέντι. You know it. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ξέρετε ήδη. Αλλά θα σύνομα να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα δράσης της Εκτελεστικής Επιτροπής που, α, που καλείται χορηγώντας ένα χρόνο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ισότητας ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες που λέγεται γενικά πρόγραμμα Στοκόλμης. Αυτό το πρόγραμμα δράσης είναι κατευθυντήρια γραμμή για την αθέτηση πολύ συγκεκριμένων μέτρων τα επόμενα πέντε χρόνια. Αν κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξή εδώ τώρα έχει αποδεχθεί από τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, των τελευταίων μηνών, ότι υπάρχει ένας χαρακτήρας επίγον για να αντιμετωπίσουν οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Ευρώπης. Καθώς επίσης πολύ καθαρές ε, ε, προσδοκίες των πολιτών ότι πρέπει να δράσουν γλίγορα και αποτελεσματικά. Α θυμηθούμε την αθέτηση του προγράμματο ε, εργασίας στις εκτελεστικές επιτροπές. Ήδη από το περιεχόμενο του καταδεικνύει ότι η εκτελεστική επιτροπή είχε όχι μόνο την πρόθεση να δράσει, αλλά δρά. Μεταξύ άλλων εστιασμένη στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει μια ατζέντα των πολιτών που θέτει τους πολίτες στο επίκεντρο, στην καρδιά της ευρωπαϊκής δράσης και το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της δικαιοσύνης και της εσωτερικής πολιτικής είναι η πρώτη στρατηγική πρωτοβουλία της νέας εκτελεστικής επιτροπής τόσο ώστε αυτό το πρόγραμμα ε, εργασίας να τεθεί σε ισχύ και ακολουθεί αυτό πολύ στενά την εντολή που δόθηκε σαν ευρύτερη φιλοσοφία από το πρόγραμμα της Στοχόλμης και λαμβάνει επίσης υπόψη τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η πρόκληση να εξασφαλίσουμε το σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών, τα ταυτόχρονα και μια εγγύηση για την ασφάλεια στην Ευρώπη, είναι αυτό που αντιμετωπίζεται εδώ σφαιρικά, θα λέγαμε και υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες που αναφέρονται που είναι ένας οδικός χάρτης για μια ελεύθερη και ασφαλή Ευρώπη. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορεί κανένας να αποχωρήσει την ασφάλεια από την ελευθερία. Είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Σχετίζονται όμως όλες με τους πολίτες και είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε οι πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρώπη. Το πρόγραμμα δράσης θα μας κατευθύνει για να καταλήξουμε σε ένα σύνολο πολύ φιλοδόξων μέτρων σε ένα τομέα στον οποίο θα ήταν πολύ ορατή η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης για τους πολίτες. Πρόκειται λοιπόν και για ένα ισχυρό μήνυμα, αυτό που συζητούσαμε προηγουμένα, που η συνθήκη της Λισαβόνας και η Ευρωπαϊκή Χάρτα Βασικών Δικαιωμάτων είναι δράσεις υπέρ των πολιτών. Επειδή όλες αυτές οι δράσεις είναι αλληλένδετες, απαραίτητες και ε, με συνέχεια στους όρους που έχουν οριστεί από συνθήκες της Αβώνης και στον, στη Χάρτα Βασικών Δικαιωμάτων, θα πρέπει να πετύχουμε την ε, πραγματοποίηση των ε, φιλοξών με αυτό το γλυγορότερο δυνατόν ευθυγραμμισμένη και με τις προσδοκίες των πολιτών. Και γι' αυτό αυτό το πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Κοινοβούλιο όχι σαν κάτι το οποίο είναι αμετάκλητο, γιατί μπορεί να υπάρξει κάτι το απρόβλεπτο και γι' αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή οπωσδήποτε αν υπάρχει κάτι το απρόβλεπτο θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμά της πρωτοβουλίας για να επιλύσει τα προβλήματα και αυτό θα είναι σημαντικό για το Βούλιο. έχουμε ε, την πρόθεση να υποβάλουμε μία προσωρινή ε, αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος Σοκόλμης το 2012 για να είμαστε σε σίγουροι εξακολουθεί το πρόγραμμα να παραμένει ευθυγραμμισμένο με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος ο Υπουργό δικαίως, αυτό το πρόγραμμα δράσης δεν αφορά μόνο το τι θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επίσης αφορά και το τι πρόκειται να κάνουν τα κράτη-μέλη. Πώς τα κράτη-μέλη θα αναλάβουν τις δικές τους πρωτοβουλίες όπου χρειάζεται η πρωτοβουλία, όπου υπάρχει επικουρικότητα, πώς τα κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εθνική τους νομοθεσία και πώς θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τη συνεργασία με τα άλλα κράτη-μέλη. Αυτό το πρόγραμμα δράσης, αγαπητοί βουλευτές, θα είναι επιτυχή στο τέλος μόνο αν όλα τα θεσμικά όργανα παίξουν το ρόλο τους. Και έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε γρήγορα στη σωστή άγουσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα τη συζήτηση με τους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων και ξεκινάμε με το ΕΛΚ για 1,5 λεπτό. Γκοράτσα Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ε, κατέθεσε έγκαιρα ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης που ε, δίνει μεγάλη σημασία, προβάλλει την εικόνα του Ευρωπαίου πολίτη. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε σε μια Ευρώπη με επίκεντρο τον πολίτη για τον πολίτη, για τον Ευρωπαίο. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραμείνει προσιλωμένη σε αυτό το όραμα όταν θα καταθέσει τις προτάσεις της για τα επόμενα πέντε χρόνια. Το πρόγραμμα λοιπόν αποτελεί μια πραγματική ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια που θα προσφέρουμε στους πολίτες ενώ παράλληλα θα σεβόμαστε τα δικαιώματά τους, τις ελευθερίες τους, ε, την ακαιρεότητα και την έννοια της, ε, του ενεργού πολίτη. Αυτό που έχει σημασία είναι να ενισχύσουμε την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Θα ήθελα επίσης να πω ότι το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει και μια στρατηγική για να καταπολεμηθεί η κακοποίηση, ο κροτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών και θα ευχόμουν αυτή η πρόταση να έχει ήδη κατατεθεί νωρίτερα. Επίσης ε, πρέπει να ενθαρρύνουμε και τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία και να διασφαλίσουμε τη διασφάνεια. Ελπίζω λοιπόν τα μέτρα να ε, παρουσιαστούν με φιλικό τρόπο. Ολοκληρώνοντας προσβλέπω στη συνεργασία με τους συναδέλφους μου στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο έτσι ώστε να προσφέρουμε πραγματικά ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης και αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Γκουενς, ε, επόμενος ομιλητής, ε, για 1,5 λεπτό. Κυρία Γκουενς. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις τεχνικής φύσεως. Βεβαίως και πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό πρέπει να πω ότι είμαστε κατά τη απογοητευμένοι γιατί ε, οι ε, φιλοδοξίες ε, που αναφέρονται σε αυτό δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε. Και γι' αυτό εμείς εκφράσαμε την δυσαρέσκειά μας με κατάθεση τροπολογιών. Υπάρχουν αρκετά σημεία στο πρόγραμμα που προβλέπουν σημαντικά ότι το 2013-2014 ήδη πρόκειται για καθυστέρηση. Και υπάρχει και άλλο ένα πρόβλημα που έχει σχέση με τις ε, διεθνείς ε, συμφωνίες, με τη συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Η συνεργασία αυτή δεν είναι απόλυτα σαφής. Παρότι έχει υπάρξει κάποια βελτίωση, παραδείγματος χάρη, ε, στις διαπραγματεύσεις για το SWIFT με τις Ηνωμένες Πολιτείες βελτιώθηκε κατά την κατάσταση, κυρίως την αντίδραση, αλλά ακόμα δεν λύθηκε το πρόβλημα. Έχουμε τη συμφωνία πλαίσιο, η οποία είναι η μόνη που προβλέπεται πιο συγκεκριμένα. Οι πολίτες τελικά. Ο πολίτης ε, δεν προβάλλεται επαρκώς ε, κάτω από το πρίσμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται σωστά. Και όσον αφορά στη μετανάστευση, αρχίσαμε τη συνεργασία, αλλά όπως σας είπα οι στόχοι δεν είναι αρκετά υψηπετής. Αυτή λοιπόν η αμοιβαιότητα απαιτεί νέες αποτελεσματικές λύσεις γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν εκρεμή προβλήματα και η ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων ε, θα πρέπει να λαμβάνει η χώρα χωρίς διακριτική μεταχείριση. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Βίμπα για 1,5 λεπτό εκ μέρους των φιλελευθέρων. Κυρία Βίμπερ, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φιλόδοξο το πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να εγκριθεί σχέδιο δράσης για να υλοποιηθεί ώστε τον πιο αποτελεσματικά. Και αποτελεσματικό δεν σημαίνει, δεν είναι μόνο να έχουμε σωστό χρονοδιάγραμμα, αλλά αποτελεσματικό σημαίνει να ε, συμβάλλει επίσης ε, στα νομοθετήματα που θα υιοθετήσουμε τα επόμενα χρόνια, μεταξύ άλλων. Για να υπάρξει μεγαλύτερη συνέπεια σε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων, περισσότερη αστυνομική συνεργασία, ε, ό,τι έχουμε κάνει δηλαδή και με την εσωτερική αγορά. Θα πρέπει άρα να αλλάξουμε την άποψη που έχουμε για τα εθνικά νομικά συστήματα, τα οποία δεν θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιούμε ή να κακοποιούμε, ώστε να έχουμε τα ελάχιστα δυνατά πρότυπα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ποινικό δίκαιο. Πρέπει να αποφύγουμε μια τέτοια προσέγγιση, θα πρέπει να έχουμε ε, περισσότερη περισσότερη ε, προστασία του πολίτη από, έναντι της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και το καθεξής. Να ασπίσουμε τα δικαιώματα των θυμάτων αλλά και των εναγόμενων. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα που να ισχύουν παντού, σε όλα τα κράτη-μέλη. Οφείλουμε να είμαστε θαραλέοι, να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες στη Eurojust, να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών μας, να νομοθετήσουμε σωστά ε, για το άσυλο. Η πολιτική μου ομάδα θα δουλέψει επικοδομητικά με την Επιτροπή, με το Συμβούλιο και ε, θα πολεμήσει για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Σαρτζεντίνη για δυόμιση λεπτά εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούγοντας ε, την Επίτροπο και το Συμβούλιο για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, ε, μου έρχονται κάποια ερωτηματικά. Τώρα τελειώνει πια σχεδόν η Ισπανική Προεδρία σε πέντε περίπου εβδομάδες και ακούσαμε στην αρχή όταν ανέλαβε η Ισπανική Προεδρία την ε, θητή αυτή να ε, εκφράζει πολλές κορώνες ε, για τη μετανάστευση για τις γυναίκες και διαρωτώ με σε αυτές τις πέντε εβδομάδες που λείπουν τι θα γίνει τελικά με συγκεκριμένες προτάσεις για αυτά τα θέματα η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έκαναν τη δουλειά τους για το άσυλο και τη μετανάστευση και περιμένουμε τώρα το Συμβούλιο να δραστηριοποιηθεί δεν είναι όπως είπε η κυρία Ρέντινγκ ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τους νόμους τους. Το Συμβούλιο είναι εκείνο που θα πρέπει να τοποθετηθεί για τη συνθήκη του Δουβλίνου, ε, της υποδοχής μεταναστών, ε, για πολλά. Εμείς περιμένουμε. Η οδηγία κατάργησης διακρίσεων ε, ψηφίστηκε σε αυτήν την Ολομέλεια και οι πράσινοι περιμένουν να μεταφραστεί στην πράξη. Και Βεβαίως ε, ισότητα και κατάργηση διακρίσεων είναι απολύτως απαραίτητες ε, που αναφέρονται στο πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης. Όμως γιατί η Επιτροπή επέλεξε να μην καταστήσει τα θέματα αυτά προτεραιότητα, προτεραιότητα στο πρόγραμμα δράσης. Είπατε ότι ο πολίτης πρέπει να μπει στο επίκεντρο συνεργασία ισότητα των φύλων, αυτά είναι τα σημαντικά. Και όσον αφορά τη Europol, πριν από τη Λισαβόνα η Europol ε, υφίστατο έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό, παρότι βέβαια ισχύει η συνθήκη τη ε, Λισαβόνα. Παραδείγματο χάρη, οι ε, αρμοδιότητε για να υπάρξουν ε, συμφωνίε συνεργασία με τρίτε χώρε. αυτό βασίζεται σε μια απόφαση βουλή πριν από κάποια χρόνια. Κυκλοφορούν φήμε ότι τώρα η Europol συζητά να συνάψει συνθήκη, συμφωνία με το Ισραήλ και ποτέ δεν ξέρει κανείς και ποιες άλλες χώρες θα μπορούσαν να υπογράψουν συμφωνίες με μας. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει ένα νέο ρόλο και καλό την Επιτροπή να δράσει ανάλογα. Η κυρία Μπιτσότο, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχουμε 160 διατάξει σε τρία χρόνια. Ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, ηχεί τουλάχιστον αυτό με την πρώτη ματιά. Όσον αφορά την ε, μετανάστευση, βέβαια τα πράγματα είναι πολύ δυσάρεστα. Ε, θα έπρεπε να προαχθούν ε, οργανισμοί και αυτό όμω πάλι δεν φτάνει. Υπάρχει μια πραγματική στρατηγική η οποία θα βασίζεται στον αγώνα κατά της λαθρομετανάστευσης στις διαφορές βορρά-νότου. Ε, να μην υπάρχουν διαφορές στα κρατημέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Να αναγνωριστεί ότι η μετανάστευση ε, δεν μπορεί να αποτελεί πηγή για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Εμείς ε, θεωρούμε ότι πάνω από το 20% των ανέργων στην Ευρώπη είναι νέοι σε μία ήπειρο με εκατομμύρια ανέργους. Λέμε ότι η Επιτροπή Μετανάστευσης πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη. Να δουλεύει συγκεκριμένα και με ρολισμά. Σήμερα η πρώτη προτεραιότητα είναι να δώσουμε εργασία στους πολίτες μας βεβαίω το να παραμένει κανείς ε, θεωρητικός αυτό δεν βοηθάει τους μετανάστευση πόσο μάλλον τους δικούς μας ανθρώπους. Τώρα, θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους μελητές Ντεμέρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μιλούμε για πάνω από 360 δράσεις σε 5 χρόνια. Θα έπρεπε λοιπόν να ασχοληθεί περισσότερο το Κοινοβούλιο το θέμα αυτό και να μπορέσουν τα μέλη να εμβαθύνουν σε κάθε μία από αυτές τις προτάσεις, το περιεχόμενό τους. Θα έπρεπε να έχει δοθεί περισσότερο χρόνο, ε, περισσότερος χρόνος. Για παράδειγμα, παρακολούθηση των διάβλων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας των τέτοιου είδους διάβλων. Η συνεργασία Europol, Eurojust ε, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος χρήση του διαδικτύου, κανονισμός Frontex, Ευρωπαϊκό ε, σύστημα Φύλαξης εξωτερικών συνόρων και καθεξής. Σας διάβασα ένα σωρό παραδείγματα και υπάρχουν άλλα τόσα. Δηλαδή, εξαιρετικά σημαντικά θέματα και θα έπρεπε να είχε ασχοληθεί το Κοινοβούλιο με, με διάφορες συνθέσεις με το θέμα αυτό. Προστασία των θυμάτων αδικημάτων. Ε, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα συνολικό μέσο για την προστασία των θυμάτων και να συμπεριληφθούν εκεί και τα θύματα της τρομοκρατίας. Είναι μια τροπολογία την οποία δεν μπόρεσα να υποβάλω για λόγους κανονιστικούς. Ειδικό μέσο για την προστασία των θυμάτων τρομοκρατίας. θα πρέπει αυτό να ήταν βασικό στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου, κυρία Ρέντιν, πείτε μου παρακαλώ, γιατί ως προς τη Europol μια απόφαση του Συμβουλίου θα αντικατασταθεί από κανονισμό ε, για τη Europol με χρονικό ορίζοντα το 2013. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπένοβα για μισή λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, στο πρόγραμμα δράσης της ε, Στοκόλμη υπάρχουν κάποιοι τομεί του οποίους ε, θα ήθελα να θίξω ε, και θα ήθελα για να προχωρήσουμε να αναφέρω πρώτα του προβληματικούς τομεί. Κατ' εμέ, προβληματικό είναι το σύνολο του συστήματος χορηγήσης ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω αυτό το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Από τη μία πλευρά έχουμε την Κομισιόν η οποία κάνει λόγο για την ανάγκη ενσωμάτωσης των μεταναστών ε, στο σύστημά μας. Από την άλλη όμως σε αυτό το πρόγραμμα δράσης ε, δεν αναφέρονται αρκετές ε, φιλοδοξίες. Μέχρι το 2014 βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία ελπίδα έτσι ώστε οι αιτήσει ασύλου να είναι ενιαίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα Υπάρχουν ε, κάποιες ε, προτάσεις ε, για την μετακίνηση των εποχικών εργαζομένων και των ετούντων άσυλο. Κάποια θέματα που δεν προβλέπονται, αν είναι πολύ σημαντικά, είναι τα καταστηλητικά μέτρα. Και κάτι άλλο. Η Κομισιόν αναφέρει ότι οι ε, αναγνωρισμένες ε, συνεργασίες, ε, οι συνεργασίες όπου συμμετέχουν και τα δύο φύλλα δεν αναφέρονται πουθενά. Αυτό όμως είναι σημαντικό και κρίμα που λείπει. Όσον αφορά τις συνεργασίες, τελειώνοντας να πω ότι το πρόγραμμα αναφέρει τις ελευθερίες των επιχειρήσεων χωρίς όμως συγκεκριμένες ρυθμίσεις και αυτό τη στιγμή που υπάρχει κρίση νομίζω ότι ε, πραγματικά εκπλήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία λάτφορτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κατάλογος των πέντε συγκεκριμένων μέτρων για το δικαίωμα του ατόμου στις ε, ποινικέ διαδικασίε σε σχέση και με το δοδικό ε, χάρτη του προγράμματο τη Δοκόλμη είναι και το πιο θετικό ε, στοιχείο τη έκθεση του όλου κειμένου γενικότερα. Και εγώ είχα δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα και ήρθα σε συμφωνία ε, με τον εκπρόσωπο της Ισπανικής Προεδρίας. Συμφωνήσαμε σήμερα το πρωί και ελπίζω να τηρηθούν αυτά που συμφωνήσαμε. Υπάρχει πρόταση της Επιτροπής και ε, συνέβαλαν πολλοί υπηρεσίες της Επιτροπής. Θέλω να ευχαριστήσω τους αρμοδίας. Τελικά καταφέρνουμε να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη για την αμοιβαία αναγνώριση. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα πράγματα τώρα είναι μερικές φορές φρικτός. Είχαμε την περίπτωση Γκάρι Μάντεν. Αν είχαμε ε, τέτοιου είδους μέτρα στο παρελθόν, κακοδικίες ε, τέτοιου βεληνικούς δεν θα είχαν λάβει χώρα. Ευχαριστώ. Κύριος Πουσούτιλ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, η κοινή εσωτερική αγορά ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τώρα αυτό το σχέδιο το οποίο είναι υπέρ του Ευρωπαίου πολίτη και πιστεύω ότι αυτό θα είναι το καινούριο μεγάλο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, το 1992 ολοκληρώθηκε η εσωτερική αγορά και υιοθετήθηκε η συνθήκη του Μάστριχτ και τότε θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η έννοια του Ευρωπαίου πολίτη. Με αυτό το σχέδιο δράσης ε, φτιάχνουμε έναν χώρο ε, όπου πραγματικά θα εφαρμοστεί στην πράξη, θα αποκτήσει και πρακτική, ουσιαστική χρειά η έννοια της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη, θα ε, πραγματικά κατοχυρώνεται το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε πλέον παράδειγμα. Θα είμαστε χώρος, ευρωπαϊκός χώρος θα είναι χώρος σύμβολο, χώρος παραδείγματος όπου πραγματικά θα διώκονται και θα τιμωρούνται αδικήματα όπως είναι ε, το εμπόριο ανθρωπίνων όντων ή η παιδοφιλία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δοθεί σημασία στην ε, έννοια αυτή και να υπάρξει απόλυτη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική σε συγκεκριμένους τομείς. Άλλωστε το σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει και χρονοδιαγράμματα, προθεσμίες, τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε για να έχει νόημα. Ευχαριστώ. Λόπεθ Αγγιλάρ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ ήμουν συνεισηγητής μαζί με τους μαζί με τον πρόεδρο Κασίνη και το μέλος Μπέρλινγκουέρ, συνεισηγητής για το ψήφισμα που υιοθετήσαμε τον περασμένο Νοέμβριο σχετικά με το πρόγραμμα δράση της Στοκχόλμης. Και θέλω να υπογραμμίσω το εξή. Τότε είχα τονίσει ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης δεν θα καθιστούσε τη ζωή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο απλή, αλλά θα καθιστούσε την λειτουργία μας πολύ πιο απαιτητική. Διότι διάφορα τα οποία περιλαμβάνονταν ε, στην αρχή δεν αντικατοπτρίζονται με συγκεκριμένο τρόπο στο σχέδιο δράση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε ποια είναι τα όρια τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Παρ' όλα αυτά, θέλω να υπογραμμίσω ότι οι παράγραφοι 148 έως και 150 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιείχαν αναφορές σε πολύ συγκεκριμένα θέματα πολύ σημαντικά από την προστασία των θυμάτων μέχρι ε, τα θεσμικά όργανα που έχουν να κάνουν με τη συνθήκη του Σέγγεν, την Eurojust, τη Frontex, τα θέματα ασύλου και το Και ε, γίνονταν αναφορά και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και στη ρήτρα της μη διάκρισης. Ε, προστασία των δεδομένων είναι κάτι το πολύ σημαντικό και ε, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως. Θα πρέπει να βρεθεί σωστή ισορροπία, το σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ της ασφάλειας αλλά και της ιδιωτικότητας, της ιδιωτικής σφαίρας. Πέντε χρόνια έχει μπροστά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εφαρμοστεί κατά γράμμα κάθε ένα από τα σημεία του προγράμματος δράσης ε, της Στοκχόλμης. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργαστεί σκληρά, να εργαστεί σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο, ώστε να ληφθούν υπόψη τα πολύ σημαντικά περιεχόμενα των παραγράφων 148 έως 150 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάζει τη διαδικασία, θα εξετάζει τη δουλειά του Συμβουλίου και της Επιτροπής και θα εφιστά την προσοχή ε, σε σημεία που πραγματικά είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γκριέσμπεκ, ένα λεπτό. Κυρία Γκριέσμπεκ, ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, αγαπητέ εκπρόσωποι του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίηση που νιώθω διότι πλέον έχουμε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης της Στοκχόλμης. Ποικίλα τα θέματα, σημαντικά θέματα, δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλα. Θα αναφερθώ σε δύο-τρία σημεία που θεωρώ ότι αξίζουν της προσοχής μας. Πολύ στενές προθεσμίες έχουμε ορίσει για την εφαρμογή όλων αυτών. Αυτό είναι το πρώτο που θα ήθελα να πω. Θα πρέπει όλοι να δράσουμε ούτως ώστε ε, τα λόγια μας να μην είναι λόγια του αέρα αλλά να ε, μεταφραστούν και στην πράξη. Για να εφαρμοστεί λοιπόν το πρόγραμμα δράσης οφείλουμε να καθορίσουμε προτεραιότητες. Η κυρία Ρέντιν αναφέρθηκε στην προστιθέμενη αξία θεωρώ ότι τονίζουμε κάποια σημεία τα οποία θεωρούμε πιο επίγοντα και θα πρέπει επομένως να επιταχύνουμε ε, ε, σε θέματα δικαστικής συνεργασίας να έχουμε ας πούμε πρόγραμμα εράσμους των δικαστών και όχι μόνο των δικαστών, όλων των νομικών επαγγελμάτων αλλά και των ε, νομικών που εργάζονται στους κόλπους των αστυνομικών αρχών. Να επιταχύνουμε λοιπόν σε θέματα δικαστικής συνεργασίας, να επιταχύνουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με το κύβερνο έγκλημα, την παιδική ε, πορνογραφία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση ε, και το, εν γέννη όλα τα αδικήματα που διαπράττονται εις βάρος των παιδιών. Ευχαριστώ κύριε Λαμπρινίδη, ένα λεπτό. Άλλη που λείπει από τα προγράμματα μετανάστευσης είναι η λέξη αλληλεγγύη. Ψηφίσαμε σήμερα για την επανεγκατάσταση ε, δικαιούχων ασύλου από τρίτε χώρε στην ευρώπη αλλά αρνείται το πρόγραμμα τη επιτροπή να προβλέψει αντίστοιχη πρόβλεψη για ε, εγκατάσταση ετούντων άσύλου από μια χώρα τη Ευρώπη στην άλλη ή χρήματα. πού πήγε η αλληλεγγύη; εκατό εκατο χιλιάδε και πάνω λαθρομετανάστε έρχονται στην ελλάδα από την τουρκία κάθε χρόνο. τι γίνεται με τη συμφωνία Ευρώπη Τουρκία για την επιστροφή των μεταναστών αυτών; καρκινοβατή και δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου στο πρόγραμμά σας. Τι γίνεται με τη συμφωνία που διαπραγματεύεται η Frontex σήμερα με την Τουρκία. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν θα αμφισβητεί άμεσα ή έμεσα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας αλλά της Ευρώπης. Συνοριακά. Και τέλος φυσικά η μεγάλη υποχρέωση αλληλεγγύης προς τους ίδιους τους μετανάστες που λέγεται ένταξη μεταναστών. Χωρίς την ένταξη μεταναστών κυρία επίτροπε δεν υπάρχει πιθανότητα 40 εκατομμύρια άνθρωποι που ήρθαν ανάμεσά μα να μπορέσουν να ζήσουν ισότιμα μαζί μα. δημιουργούμε πιθανέ ορολογιακέ βόμβε. χρειάζονται προγράμματα χρήματα και δεν τα έχει αυτή τη στιγμή η επιτροπή. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αουράτζι για ένα λεπτό. Έχω την εντύπωση ότι στην Ευρώπη χωρίς σύνορα με όλο και περισσότερα δείγματα υπερεθνικής εγκληματικότητας, δηλαδή εγκληματικότητας που ξεπερνά τα σύνορα ενός κράτους μέλους, τότε θα πρέπει να αυξηθούν οι απαντήσεις που δίδονται σε υπερεθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερες φιλοδοξίες ε, για τα θέματα ε, του Ευρωπαίου Εισαγγελέα ε, για θέματα εμβάθυσης της αστυνομικής συνεργασίας, της δικαστικής συνεργασίας, της ενοποίησης του ε, δικαστικού ποινικού δικαίου. Για όλα αυτά αυτούς τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Υπάρχουν πολλές εθνικές αντιστάσεις που δεν έχουν καμφθεί ακόμα. Επιμένω, το Συμβούλιο πρέπει πια να αφήσει κατά μέρο την κυριαρχική διάθεση των κρατών μελών, να ενοποιήσουμε τα, ε, την ποινική δικονομία που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος για να δώσουμε υπερεθνική απάντηση σε υπερεθνικά προβλήματα. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε τη διαδικασία Catch Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανώς ε, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή που προσφέρει το πρόγραμμα της Οκχόλμης ε, ε, πολλές δράσεις που πρόκειται και σκοπεύει η Επιτροπή να αναλάβει σε τομείς όπως είναι η ελευθερία και η δικαιοσύνη και η ασφάλεια. Βέβαια υπάρχει και το θέμα της συνεργασίας ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ανάμεσα στα ίδια τα κράτη-μέλη. Ε, αυτό είναι ένα ε, θέμα πολύ σημαντικό και πρέπει να αναζητηθούν τα πραγματικά εργαλεία συνεργασίας. Έχουμε μεταναστευτικές ροές, ε, έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα κρατούνται σε υπερσυνοστισμένες φυλακές. Άτομα τα οποία έχουν μπει μέσα σε αυτό το ε, τούνελ της, ε, των ναρκωτικών. Έχουμε το οργανωμένο έγκλημα ε, σε επίπεδο υπερεθνικό. Όλα αυτά απαιτούν να υπάρχει πραγματική συνεργασία. Και αυτή η πρόκληση είναι εκείνη που αντιμετωπίζει το δικό μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο βεβαίως καλείται να θέσει τα θέματα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως και απέναντι στα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε πολύ. Μπάτεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία ε, Πρόεδρε. Η κυρία ε, Λατφόρτ είπε ότι ανησυχεί για τις ε, κακοδικίες ε, κυρίως όσον αφορά τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για δύο συγκεκριμένους ανθρώπους. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι από μόνο του μία κακοδικία. Έγινε, απορρίφθηκε ε, η έκδοση ατόμων καθαρά και μόνο για γραφειοκρατικούς λόγους. Τα βρετανικά δικαστήρια έχουν περιοριστεί στο να ε, προστατεύουν τους πολίτες τους κυρίως όταν εκδίδονται σε τρίτες χώρες. Εγώ βρισκόμουν στο εφετείο στην περίπτωση Αντιουσίμιου όπου δύο δικηγόροι δεν μπόρεσαν να παρεμποδίσουν την έκδοση του κυρίου Σίμιου παρότι όλοι στο δικαστήριο γνώριζαν ότι ε, οι ενδείξεις και οι αποδείξεις ήταν ανύπαρκτες ή ε, και φτιαγμένες από την αστυνομία. Αυτό όμως δεν είναι το θέμα. Η αστυνομία δεν θα έπρεπε να έχει δικαίωμα να ε, παρεμβαίνει σε αυτή την περίπτωση η Σάρα Λάτφορντ και άλλοι μπορεί να χύνουν τώρα κροκοδίλια δάκρυα, αλλά ε, α μην ξεχνάμε ότι αυτοί φέρνουν την ευθύνη για την αθλειότητα ε, που έχει προκληθεί. Ο κύριο Παπα-Νικολάου για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, με ικανοποίηση ψηφίσαμε στο πρόγραμμα της στοκχόλμης τις διατάξεις που αναφέρονται στην αλληλεγγύη για τα θέματα μετανάστευσης και για τα θέματα αντιμετώπισης τη παράνομη μετανάστευση. Ε, διαβάζω στο πρόγραμμα δράσης ότι το 2011 θα δημιουργηθεί, το, ε, θα δημιουργηθεί ε, ένας μηχανισμός από την Επιτροπή που θα αξιολογεί τα εθνικά συστήματα ασύλου προκειμένου να μπορέσει να συνδράμει καλύτερα τα κράτη-μέλη σε σχέση με τις δυνατότητες που το καθένα έχει και τις ανάγκες που υπάρχουν. Παράλληλα, σήμερα δώσαμε το πράσινο φως στο Κοινοβούλιο μα στην έναρξη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου στη Μάλτα το ερώτημα είναι συγκεκριμένο θα έχει σχέση η ευρωπαϊκή υπηρεσία ασύλου με αυτόν τον μηχανισμό και στα πλαίσια αυτού του μηχανισμού και της αξιολόγησης που θα γίνει προβλέπετε πρόγραμμα εσωτερικής επανεγκατάστασης προσφύγων προκειμένου να εξομαλυθούν οι ανισότητες της πιέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη μέλη. ευχαριστώ πολύ. Eh, Τελευταία παρέμβαση Μακοβέι, για ένα λεπτό. Θα ήθελα να αναφερθώ στο μηχανισμό αξιολόγησης διαφθορά στα κράτη-μέλη. Ένας μηχανισμός που προβλέπεται στο πρόγραμμα δράση. Έχουμε μία απόφαση του Συμβουλίου ε, σχετικά με το πρόγραμμα τη Στοκόλμη που αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Έχουμε και το πρόγραμμα τη Επιτροπή για την εφαρμογή του προγράμματο τη Στοκόλμη. Και τα δύο προγράμματα αναφέρονται στην αξιολόγηση των προσπαθειών κατά τη διαφθορά στα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευση από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να λειτουργήσει ένα τέτοιο μηχανισμό. Το λέω αυτό γιατί γνωρίζουμε Ελπίζουμε όλοι μας ότι μέχρι τώρα οι προσπάθειες των κρατών μελών δεν τελεσφόρησαν. Και όσον αφορά την καταλεκτική ημερομηνία για την ανακοίνωση περί διαφθοράς στο πρόγραμμα δράσης, στο μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, καταληκτική ημερομηνία είναι το 2011. Ίσως θα ήταν καλύτερα άμεσα να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αντιμετώπισης διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, η διαφθορά και αυτή η οικονομική κρίση, άρα δηλαδή μέτρα για να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα ε, θα δώσω το λόγο ε, στον ε, κύριο Λόπες Καρίντο για να μιλήσει εξ ονόματος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα η ουσία της συζήτησης για τον χώρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης, Ασφάλειας και Ελευθερίας έγκυται σε αυτό το οποίο είπε ο, το μέλος Μπουσούτιλ, ο οποίος μίλησε για την έννοια της ευρωπαϊκής ηθαγένειας, για την έννοια του Ευρωπαίου πολίτη. Αυτή τη στιγμή αυτό προσπαθούμε να χτίσουμε. Ε, πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτή την έννοια και σίγουρα ε, αυτό ήταν ένας από τους άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκε η Ισπανική Προεδρία και είναι ένας από τους άξονες της μελλοντική πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, είχαμε και την τοποθέτηση Αργεντίνη σε σχέση με τα επιτεύγματα της Ισπανικής Προεδρίας για το θέμα αυτό και για το τι προβλέπετε για το μέλλον. Σας ευχαριστώ για την άμεση ερώτησή σας με ρωτήσετε ξεκάθαρα τι έχουμε κάνει για το θέμα αυτό και θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Μιλούμε για τα δικαιώματα, για τις ελευθερίες, για έναν χώρο ασφάλειας, δικαιοσύνης, για το καθεστώς του Ευρωπαίου πολίτη στον 21ο αιώνα. Ως προς τις ελευθερίες λοιπόν, έχουμε την προσχώρηση στη Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν μία από τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας και θα εγκριθεί αύριο. Το συζητήσαμε προηγουμένως. Επίσης, σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να μιλήσουμε για την οδηγία για τις εγγυήσει ως προς τη σωστή τήρηση των δικαστικών διαδικασιών ε, και την άσκηση των εκάστοτε διώξεων. Έχουμε την οδηγία για τη μη διάκριση και περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σε γενικές γραμμές για την διάκριση. Η οδηγία αυτή είναι εξαιρετικά φιλόδοξη και εξαιρετικά σημαντική. Τη στηρίζει η Ισπανική Προεδρία και περιμένουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως προς τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα θύματα, ανησυχία, μέρημνα, της Ισπανικής Προεδρίας ήταν η προστασία των θυμάτων και ειδικότερα των θυμάτων αδικημάτων βίας που έχουν να κάνουν ε, με τα δύο φύλλα. Έχουμε την οδηγία ε, για την καταπολέμηση της σεξουαλικής ε, παρενόχλησης και εκμετάλλευσης. Αυτά θα εγκριθούν τον Ιούνιο. Δουλεύουμε πάνω στην νομοθετική πρωτοβουλία αυτή για να καταπολεμηθούν ε, τα εγκλήματα και η βία που έχει να κάνει με τα δύο φύλλα. Ουσιαστικά έτσι θα κατοχυρώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ε, προστασία και την μείωση του αριθμού των θυμάτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Έχουμε και μία ενιαία τηλεφωνική γραμμή ε, την οποία μπορούν να καλέσουν τα θύματα και να λάβουν βοήθεια εγκρίναμε τη στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια στο Συμβούλιο του Μαρτίου, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου. Εγκρίναμε τη σύσταση ε, της ε, Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας. Προχωρούν και δρομολογούνται συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ για θέματα ασφαλείας. Έχουμε τη δήλωση του Τολέδο ε, και τη δήλωση για το θέμα SWIFT, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία με τη ΣΥΠΑ το γρηγορότερο δυνατό. Από εκεί και πέρα. Έχουμε επίσης ε, δουλέψει για μια συμφωνία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, συνεργασία ε, σε θέματα αστικού δικαίου, το ΡΟΜΗ 3. Έχουμε προχωρήσει το ΡΟΜΗ 3. Σε θέματα ασύλου που αναφέρθηκαν πολύ για τα θέματα αυτά. Η Ισπανική Προεδρία όφιλε να κάνει την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Και το κάνει αυτό και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση προγράμματος για την επιστροφή μη συνοδευόμενων ανηλίκων. Ε, έχουμε και τη Frontex και ασχολούμαστε, δουλεύουμε πάνω σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους πρόσφυγες και την εγκατάσταση αυτών ή τον επαναπατρισμό αυτών, αναλόγως με τη χώρα. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους πρόσφυγες και θεωρούμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί, θα έχει συσταθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο αυτό το 2011. Υπάρχει και η έκθεση Ταβάρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα πρέπει να εγκριθεί και έχουμε δρομολογήσει διάφορες άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες για θέματα μετανάστευσης. Θέλω να σας υπενθυμίσω και τη συζήτηση στην οποία συμμετείχε με πολύ επικοδομητικό τρόπο η Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα η Επίτροπος Ρέντιν για, την, ε, για το αξίωμα, για το θεσμό του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα, κάτι που προβλέπεται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα πρέπει λοιπόν σε μια πρώτη φάση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το πολύ επίκαιρο στους καιρούς τους χαλεπούς που διανύουμε. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να είμαστε σε θέση να ασκούμε διώξεις για αδικήματα που ξεπερνούν τα σύνορα αμυγός του εκάστοτε κράτους μέλους. Είναι μια συζήτηση την οποία έχει προωθήσει και αυτή η Ισπανική Προεδρία. Σας ανέφερα έτσι επιγραμματικά διάφορα σχέδια τα οποία ξεκίνησαν, συνεχίστηκαν ή ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας και θεωρούμε ότι είναι ζωτική σημασία να αποκτήσουμε πολύ περισσότερη αξιοπιστία και πραγματικά να φανεί ότι είμαστε μια Ευρώπη ανοιχτή αλλά και ασφαλής η οποία προστατεύει ε, τους πολίτες της. ισπανικη προεδρια και θεωρουμε οτι ειναι ζωτικη σημασια να αποκτησουμε πολυ περισσοτερη αξιοπιστια και πραγματικα να φανει οτι ειμαστε μια ευρωπη ανοιχτη αλλα και ασφαλης η οποια προστατευει τους πολιτες της αλλωστε ε, θα συνεχιστεί το έργο με τις ε, επόμενες προεδρίες Έχουμε ε, το Βέλγιο και την Ουγγαρία και συνεργαζόμαστε ε, με αυτές αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δοθεί συνέχεια σε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Επίτροπος κυρία Ρέντιν. Όλοι μιλάνε για το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης. Είναι σαν ένα ε, χριστουγεννιάτικο δέντρο με συνδυασμένο με εκατοντάδες ευχές χιλιάδες ευχές εγώ όμως θα ήθελα να μιλήσουν όλοι για την πραγματικότητα αυτές οι χριστουγεννιάτικες ευχές πώς αντιμετωπίστηκαν πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας και κλεισμένων των θυρών αντιμετωπίστηκαν χωρίς να ληφθούν επαρκώς υπόψη οι πολίτες το ότι επιθυμούν, εύχονται και αναμένουν. Στον τρίτο πυλώνα, οι Υπουργοί Εσωτερικών δεν ρώτησαν δεν απευθύνονται ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είχε καμία δυνατότητα παρέμβασης. Εκεί λοιπόν βρισκόμαστε, από εκεί ξεκινάμε, από μια απαράδεκτη κατάσταση, όπου οι ελάχιστες, οι αποφάσεις δεμήνυμες, ούτε καν αυτές εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, όπου οι πολίτες δεν είχαν καν τα μέσα, τα εργαλεία να καταφύγουν στο δικαστήριο, να διαμαρτυρηθούν και να δικαιωθούν. Ευτυχώς λοιπόν τώρα έχουμε τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Δεν υπάρχει πλέον τρίτος πυλώνας. Υπάρχουν οι προτάσεις της Επιτροπής, ε, η συναπόφαση, η εφαρμογή σε επίπεδο κράτους μέλους, ε, ο έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όμως αυτό σημαίνει παράλληλα ότι τα πράγματα πλέον ε, δεν γίνονται αυτόματα. Έχουμε κανόνες, οι προτάσεις ε, πρέπει να ακολουθούν την πεπατημένη, ε, μια πεπατημένη που ζητήσατε εσείς αγαπητοί ευρωβουλευτές, τη ζητήσατε από την Επιτροπή να την εφαρμόζει στη δουλειά της. Που σημαίνει, πρώτον, εμβριθείς ανάλυση του τι είναι εφικτό, τι είναι καλό, τι προσφέρει υπεραξία. Δεύτερον, δημόσιες διαβουλεύσεις έτσι ώστε να καθίσατε σαφές ότι οι ιδέες που εκφράζονται θα γίνονται ή γίνονται αποδεκτές ή μήπως απορρίπτονται από την κοινωνία των πολιτών, από τους βιομηχανικούς κύκλους, από τα κράτη-μέλη, από τα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία και αυτά τώρα είναι πλέον παίκτη σε αυτό το σκηνικό και είναι εκείνα ε, τα οποία περνάνε από το τεστ της επικουρικότητας. Κατόπιν, αξιολόγηση των ε, επιπτώσεων για να γνωρίζουμε κατά πόσο αυτά που κάνουμε είναι σωστά και μόνο αφού γίνουν όλα αυτά, μόνο τότε θα ακολουθεί η τελική απόφαση από πλευράς Κομισιόν. Αν θέλετε λοιπόν η Κομισιόν να κάνει αυτό που έκανε τα τελευταία χρόνια, μπορείτε να μου το πείτε. Εγώ θα έρχομαι εδώ ε, κάθε εβδομάδα με μία πρόταση. Και ξέρετε τι θα γίνεται με αυτές τις προτάσεις. Αυτές ε, πρώτα απ' όλα και πολύ σωστά θα μπλοκάρονται στα εθνικά κοινοβούλια γιατί πλέον πρέπει να εμφανιζόμεθα με σοβαρό τρόπο, με σοβαρές προτάσεις που θα βασίζονται σε ε, παραδοχές νομικά τεκμηριωμένες ότι αυτά που κάνουμε είναι εφικτά. Και αφού γίνουν όλα αυτά, μετά να δούμε κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν στα κράτη-μέλη. Εγώ δεν επιθυμώ η πρώτη πρόταση που θα καταθέσουμε να αμφισβητηθεί τόσο στο δικαστήριο στο Λουξεμβούργο όσο και σε αυτό στο Στρασβούργο. Θα ήθελα λοιπόν όλοι μας να ακολουθήσουμε ένα δρόμο όπου ο πολίτης θα κατανοεί ότι η προστιθέμενη αξία που προκύπτει εδώ τον ωφελεί πρακτικά. Βεβαίως και ως ε, αρμόδια Επίτροπος για τις υποθέσεις των γυναικών άκουσα το Κοινοβούλιο να μας επισημαίνει τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε πάνω απ' όλα οι γυναίκες σε όλα τα κράτη-μέλη να έχουν τη νομική κατοχήρωση ότι όταν ή αν έχουν ποτέ πρόβλημα ε, βίας να δικαιωθούν. Να μην ε, ε, ζήσουν το δράμα του, να μην έχουν που να στραφούν. Εδώ λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε και υπάρχουν εκατοντάδες μέτρων τα οποία πρέπει να κατατεθούν πλέον με σαφή τρόπο να προσαρμοστούν σε αυτά που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, να μετατραπούν σε διατάξεις νομοθετικές. Μιλάμε για εκατοντάδες μέτρα τα οποία όμως δεν λειτουργούν στην πράξη. Η κυρία Λάτφορτ αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Βεβαίως και ε, δεν υλοποιείται στα κράτη-μέλη, διότι η όλη υποδομή η αμοιβαία αναγνώριση και η αμοιβαία εμπιστοσύνη στην οποία εδράζει η αμοιβαία αναγνώριση, δυστυχώς δεν υπάρχει, συνάδελφοι. Όλα αυτά δεν μπορεί να γίνουν αν δεν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ με εντολή να επιβάλλω την ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη στον εγκέφαλο των δικαστών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όχι έτσι πρέπει να οικοδομήσουμε αυτή την αμοιβαία εμπιστοσύνη, να την οικοδομήσουμε μέσα από νομοθετικά μέτρα και άλλα τα οποία θα συμβάλλουν στο να έρθουν στην επιφάνεια τα δικαιώματα των πολιτών σε όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι ώστε και οι δικαστές να εφαρμόζουν ε, τους κανόνες. Και προχωράμε πολύ γρήγορα σε αυτό ή ο συνάδελφος δεν είναι πια εδώ, αλλά το πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση της βίας εις βάρος των γυναικών. Το 2011 θα έχουμε ένα κείμενο που θα αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων. Κάθε είδους. Για μένα δεν υπάρχουν ε, κατηγορίες θυμάτων όλα τα θύματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Βεβαίως και ασχοληθήκαμε με την προστασία των δεδομένων. Εσείς δυστυχώς στο Κοινοβούλιο είπατε όχι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν τα πράγματα πριν τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Δεν θα συνεχίσουμε πια με αυτόν τον τρόπο. Και ναι, πρόεδρε της Επιτροπής, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι δικοί σας αλλά και οι άλλες επιτροπές εντάσσονται πλήρως ε, στον τρόπο με τον οποίο προχωράμε. Ε, πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολλά μαζί. Υπάρχουν ε, τεχνικής φύσεως θέματα, πολλά, ε, τα οποία θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις ε, κοινωνίες μας και κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες τι ακριβώς κάνουμε. Γιατί και αυτό είναι τμήμα του όλου. Και δεν είναι και το ευκολότερο. Πράγματι, πρέπει να λάβουμε μέτρα. Παραδείγματος χάρη για την ε, παράνομη μετανάστευση και για τη χορήγηση ασύλου. Η συναδελφό μου, κυρία Σεσίλια Μάλστρομ, ε, κατέθεσε πολύ συγκεκριμένε προτάσεις για την λαθρομετανάστευση, για τους ελέγχου ε, στα σύνορα. Πράγματι θα ήταν σημαντικό το Κοινοβούλιο να μπορούσε από κοινού με το Συμβούλιο να εγκρίνει τις ε, κατατεθειμένες προτάσεις για το άσυλο, για το πρόγραμμα κοινή εγκατάστασης, για την αμοιβαία αναγνώριση και για το μόλις ε, εγκριθέν πρόγραμμα δράσης σχετικά με τους ασυνόδευτους ανήλικους. Υπάρχουν πάρα πολλά εντογίγνεσθε και το θέμα δεν είναι ποιος θα κάνει τι. Γιατί ορισμένα πράγματα απλά δεν μπορεί κανείς να τα κάνει. Ας αναφέρω ένα παράδειγμα. Εσείς ζητάτε την οδηγία κατάργησης διακρίσεων οδηγία κατάργησης διακρίσεων, λυπάμαι πάρα πολύ που θα το πω, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ομόφωνα και αυτό δυστυχώς μπλοκάρεται στο Συμβούλιο. Τι να κάνω κι εγώ. Όχι εγώ, ε, πριν από μένα η Επιτροπή είχε καταθέσει την ε, ε, κατάργηση διακριτικών μεταχειρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν με αυτούς θα πρέπει να μιλήσετε, με αυτούς που τον μπλόκαραν, με το Συμβούλιο. τώρα, ε, ζευγάρια ιδίου φίλου, Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι πρόνοιες της επικουρικότητας, η αρμοδιότητα των κρατών μελών είναι εκείνη που καλείται να ρυθμιστεί το θέμα της ε, αντιμετώπισης ε, των ζευγαριών ιδίων φίλων, Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητες για τη διασυνοριακή μεταχείρισή του, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά της Γαλλίας, της Ιταλίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Ελλάδας και Λουξεμβούργου. Αυτό πρέπει να το πράξουν τα ίδια τα κρατημέλη. Βλέπω ότι ή μπορώ να δω ότι δεν θα υπάρχει αυτό που αφορά εμένα είναι να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση εις βάρος των ανθρώπων αυτών, κυρίως όσον αφορά στην κινητικότητά τους, δηλαδή όταν φεύγουν από ένα κράτος μέλος. Και εμείς αυτό αρχίσαμε να το κάνουμε. Αρχίσαμε να λέμε ότι όσον αφορά την κινητικότητα, τα δικαιώματα των πολιτών, τη συνεργασία ανάμεσα στα νομικά συστήματα, ανάμεσα ή, ε, για να το πω αλλιώς, όσον αφορά στην κατάργηση των συνόρων που εξακολουθούν να υπάρχουν σε αυτήν την ενιαία αγορά, που λυπάμαι πάρα πολύ που θα το πω, δεν είναι ε, ενιαία, δεν είναι κοινή αγορά όταν πρόκειται για τον πολίτη. Διάβασα την έκθεση του κυρίου Μόντι και εκεί στην έκθεση αυτή υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που επισημαίνουν προς τα που πρέπει να μετακινηθούμε. Και ξέρετε για μένα ποιο είναι το Ευαγγελιό μου. Η έκθεση η οποία καταρτίστηκε από ένα συνάδελφό σας. Έκθεση η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στην ελεύθερη μετακίνηση πολιτών και όλα τα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν. Αυτό λοιπόν που προτείνω εγώ σε εσά είναι να πάρετε αυτά τα προβλήματα ένα προς ένα και να τα λύσετε κι εσείς όλα αυτά ένα προς ένα όταν εγώ καταθέτω μία πρόταση και, έχετε, και βλέπετε ποια θα είναι η εξέλιξη, γιατί βέβαια έχετε πάρα πολλές ε, προτάσεις ε, μπροστά σας που ε, θα πρέπει να δουλεύετε και τη νύχτα. Δεν ξέρω αν αυτό επιτρέπεται με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και την, εργα... την νυχτερινή εργασία ανθρώπων, αλλά εγώ σας καλό να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα, γιατί εμεί θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι να απειληθούν όλα αυτά. Και δεν μπορώ να το κάνω αυτό μόνη μου. Χρειάζομαι τη βοήθειά σα. Ξέρω που θέλω να βαδίσω, αλλά βοηθήστε με να λύσω το ένα θέμα μετά το άλλο, ακόμα και αν πρόκειται να είναι ένα θέμα κάθε εβδομάδα, αυτά τα θέματα θα έρθουν στο τραπέζι σας. Εγώ με μεγάλη μου χαρά ε, να έρχομαι στις επιτροπές σας όσο συχνά επιθυμείτε και με καλείτε κύριε Πρόεδρε και θα τα ε, συζητάμε αυτά σε πέντε, μετά από πέντε χρόνια θα την έχουμε αλλάξει αυτήν την Ήπειρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, πολύ. ευχαριστώ πολύ. Κλείνει η συζήτηση εδώ.